είναι η έκθεση Λουίς Τεγκράντες Πασκουάλ για τη ρήμανση την προερχόμενη από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για τις παραβάσεις. Πρώτος ομιλητής ο ίδιος Τεγκράντες Τε Πασκουάλ, τέσσερα λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, κύριε Ταγιάννη, Επίτροπε, εκπρόσωποι του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εγώ έχω μια εξαιρετική έκθεση στο τέλος της θητείας μας που αφορά την ρήπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων ποινικών μεταξύ άλλων για τις παραβάσεις. Ελπίζω ότι η έκθεση θα τύχει της υποστήριξής σας. Ελπίζουμε ότι επειδή επιδεύτηκε συμφωνία αύριο θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία στα πλαίσια της πρώτης ανάγνωσης. Στη φάση της διαπραγμάτευσης συμφωνήσανε τα τρία κοινωτικά όργανα δεδομένου ότι υπάρχει μεταξύ όλων η ιδέα ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε τις μεγάλες, ε, τα μεγάλα δικαιώματα που γίνονται κατά της προστασίας του περιβάλλοντος. Θα πρέπει η, να σας πω ότι το ε, γεγονός ότι μπορεί να επιβάλλει κάποιες κυρώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν οφείλεται σε νέα αλλά θα πρέπει να γίνει ε, ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτής της ε, προβληματικής που είναι οι παράνομες απορρίψεις ρηπογόνων ουσιών Υπάρχουν γενικοί κανονισμοί, η σύμβαση Μαρπόλ 73-78 που αφορούν αυτά τα θέματα, αλλά βλέπουμε ότι τα, οι παρόντες ε, κανονισμοί και η παρούσα ε, νομοθεσία δεν είναι αποτρεπτική. Για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε τέτοιου είδους πρακτικές, βλέπουμε ότι κάποιοι στην πράξη παρανόμως ε, και επί τούτης ρηπαίνουν, διότι είναι πιο φθηνά να πληρώσει κανείς ένα πρόσωπο πρόστιμο παρά να ακολουθήσει όλους τους κανόνες για να μην ρηπάνει. Με την εισαγωγή κυρώσεων ποινικών εκτός από τις διοικητικές αυτό το οποίο θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να αποτρέψει οποιαδήποτε παραβίαση σε οποιοδήποτε δυνατό υπαντή. Στα πλαίσια της ε, Προεδρίας της ε, Τσεχικής θα πρέπει να πω ότι ε, έγιναν μεγάλες προσπάθειες για να μπορέσει να υπάρχει μεταρρύθμιση και αναθεώρηση της οδηγίας που θα σέβεται πλήρως την αρχή της επικουρικότητας. Η... Στην οδηγία αναφέρονται οι τρόποι με το οποίο μπορεί κανείς, ο κανένας να ενεργήσει, ενώ η πλήρης αρμοδιότητα για την εφαρμογή τέτοιου είδους αποφάσεων, εκτός από την κοινότητα που, ε, δρά επικουρικά, είναι στα κράτη-μέλη. Μέχρι τώρα αυτό το οποίο μπορέσαμε να κάνουμε είναι να μην επαναλάβουμε αυτά τα οποία είχαν γίνει στα πλαίσια της ε, οδηγίας και του πλαισίου οδηγίας του παρελθόντων, αλλά να δώσουμε μία νέα νομική βάση για να δώσουμε την δυνατότητα στον κοινοτικό ε, νόμοθέτη να μπορέσει να προτείνει κάποια μέτρα στα πλαίσια του κοινοτικού δικαίου εκτός από τα διάφορα εθνικά δίκαια. Αυτό είναι κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ε, θαλάσσιες μεταφορές και για την προστασία του περιβάλλοντος. Ξέρουμε ότι πολλές φορές οι διάφορες παράνομες απορρίψεις ρηπογόνων ουσιών ίσονος σημασία όπως λέγονται είναι κάτι το οποίο αθρηστικά μπορεί να προκαλέσει ένα μεγάλο πρόβλημα στις θάλασσες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τους και όλους οι ηγητές οι οποίοι με βοήθησαν στο έργο μου που με υποστήριξε στις διαπραγματεύσεις που έκανα με τα άλλα δύο κινητικά έργανα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τις επιτροπές που γνωμοδότησαν. Τελικά πρέπει να πω ότι καταλήξαμε σε λύση συμβαστική για τη θέση ε, ισχύ της οδηγίας που θα γίνει τους επόμενους 12 μήνες. Σήμερα νομίζω ότι όλοι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι αγαπητοί συνάδελφοι διότι έτσι και με την υιοθέτηση του τρίτου ε, πακέτου στις αρχές ε, Μαρτίου κάνουμε κάτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές. Σας ευχαριστώ. Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ευαρεσκιά της για το αποτέλεσμα στο οποίο φτάνουμε και το οποίο θα μας οδηγήσει στην υιοθέτηση μιας νέας οδηγίας η οποία να τροποποιεί την παλαιότερη. Έτσι θα καλυφθεί το νομικό κενό το οποίο δημιουργήθηκε μετά από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου η οποία ακυρώνει την, την απόφαση πλαίσιο 205-667 η οποία καθορίζει την μορφή των κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων που προκαλούν ρήπανση από τα πλοία. Μα επιτρέπει η νέα οδηγία να καταπολεμήσουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τη μόλυνση στο θαλάσσιο περιβάλλον. Είναι μια ολοκλήρωση θα έλεγα του τρίτου πακέτου για την ασφάλεια στη θάλασσα που υπεψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο παλαιότερα, στην προηγούμενη μάλλον ολομέλειά του. Στα πλαίσια αυτής της συμβιβαστικής πρότασης, η οποία βρίσκεται υπό συζήτηση, έχουμε να κάνουμε με κάποιες αλλαγές από την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρ' όλα αυτά η πρότασή σας κρατά τα βασικά χαρακτηριστικά της αρχικής μας πρότασης, τον ποινικό χαρακτήρα, δηλαδή των μέσων που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την επιβολή των κυρώσεων. Θα πρέπει να διώκονται όλοι οι υπεύθυνοι και τα νομικά φυσικά πρόσωπα. Γι' αυτό και ακριβώς υποστηρίζουμε τη συγκεκριμένη πρόταση αν και κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στις πράξεις ελάσσονος σημασίας με αυτές οι οποίες είναι ιδιαιτέρως σημαντικές και κρίσιμες. Υπάρχει θέμα παραβάσεων που δεν οδηγούν στην μόλυνση των υδάτων των θαλασσίων οπότε εκεί δεν θα υπάρχει χρήση των κυρώσεων. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να απαγορεύονται αυτού του είδους οι μολύνσεις οι οποίες, ή μάλλον αυτές οι ενέργειες οι οποίες μπορεί μακροπρόθεσμα να δημιουργήσουν προβλήματα στο θαλάσσιο περιβάλλον εφόσον μάλιστα είναι κάτι το οποίο γίνεται επαναληπτικά και εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσπάθεια την οποία κάνατε. Ευχαριστώ και τις υπηρεσίες των γραμματιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι όλοι είμαστε ικανοποιημένοι σήμερα και να στείλουμε ένα μήνυμα υπέρ της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ευχαριστώ κύριο Δόκτωρ Ματσάκης. Ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το νομικό πλαίσιο μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου οδήγησε αυτή την οδηγία προς συζήτηση αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να δούμε ότι αυτή η πολύ σημαντική οδηγία έχει καθυστερήσει σήμερα όσον αφορά την υλοποίησή τη, κάτι το οποίο έχει πολύ αρνητικέ συνέπειες για το θαλάσσιο περιβάλλον. Θα πρέπει όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία να συνειδητοποιήσουν τι αρνητικέ συνέπειε που να έχει περαιτέρω καθυστέρηση για το μέλλον του θαλασσίου περιβάλλοντος. Το συντομότερο δυνατόν λοιπόν θα πρέπει να εφαρμοστεί η οδηγία αυτή, καθότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα σταματήσουν όλες αυτές οι παράνομες απορρίψεις ρηπογόνων ουσιών από πλοία και θα αρχίσει να ελέγχεται αυτή η παράνομη δραστηριότητα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να κρατήσουμε το θαλάσσιο περιβάλλον καθαρό. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον εισηγητή για την εξαιρετική του εργασία. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Λίχτενμπεργκερ, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ρήπανση των θαλασσών είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα όλους μας μόνο και εφόσον υπάρχει ένα θεαματικό γεγονός, μια ρήπανση η οποία βρίσκεται στην επικαιρότητα και η οποία προκαλεί το ενδιαφέρον όλων μας. Μόνο τότε συζητάμε τα θέματα αυτά. Οι συνεχείς παραβιάσεις, οι συνεχείς παρανομίες οι οποίες επιβαρύνουν καθημερινά όχι μόνο τις θάλασσές μας αλλά και τις ακτές θα πρέπει να ληφθούν πολύ πιο σοβαρά υπόψη από όλους μας συχνά συζητώντας με τους συναδέλφους πιο πόσο λίγη ευαισθητοποίηση υπάρχει. Ευχαριστώ λοιπόν ιδιαίτερα τους συναδέλφους που οδήγησαν το θέμα αυτό στη σημερινή συζήτηση. Εγώ δεν ανήκω σε μια παράκτια περιοχή. Παρόλα αυτά θεωρώ ότι η απαράδεκτη ρήπανση στις ευρωπαϊκές θάλασσες είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολεί όλους έτσι ώστε οι αρχές του δεύτερου και τρίτου θαλάσσιου πακέτου να ενσωματωθούν στην δράση μας, κάτι το οποίο πραγματικά είναι επίγον. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιαζεμπόφσκι, δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, η ομάδα του ΕΛΚ βεβαίως και στηρίζει αυτήν την πρόταση τροποποίησης της οδηγίας ιδιαίτερα για περιπτώσεις πολλαπλών ε, ρηπάνσεων. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την προσπάθεια της Επιτροπής και της προσπάθειες αυτές που οδήγησαν σε αυτόν τον συμβιβασμό, στον οποίο πολύ δύσκολα θα είχαμε φτάσει χωρίς την βοήθεια της Επιτροπής. Η απόφαση του 2005 και του 2007 του Ευρωπαϊκού Δικοστηρίου σαφώς και έθεσαν στο προσκήνιο το θέμα των αυστηρότερων κυρώσεων, των ποινικών κυρώσεων θα πρέπει να έχουν αυτές οι παράνομες πράξεις. Χρειαζόμαστε αυστηρότερους κανόνες έτσι ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τις θάλασσές μας από συμπεριφορές απαράδεκτες πληρωμάτων, πλειοκτητών που πολλές φορές θεωρούν ότι οι κανόνες και η νομοθεσία που υπάρχει και ισχύει σήμερα στην Ευρώπη δεν είναι αρκετά αυστηρές και αποτρεπτικές. Ευχαριστώ λοιπόν ιδιαίτερα τον εισηγητή, ιδιαίτερα για όλες αυτές τις προτάσεις, έτσι όπως αποφασίστηκαν και συμφωνήθηκαν. Είναι πολύ πιο δύσκολο σήμερα να υπάρξουν παραβιάσεις. Η ρήπανση σήμερα αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο. Υπάρχει ταξινόμηση των ε, παραβιάσεων αυτών ανάλογα με τη σοβαρότητα, ανάλογα με τις ρηπογόνες ουσίες και ανάλογα με το αν πρόκειται για μία πρώτη φορά ή αν πρόκειται για κατεπανάληψη παραβίαση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης και το Συμβούλιο και την Επιτροπή για την επικοδομητική του στάση. Ζητώ από όλα τα κράτη-μέλη, τα οποία έχουν δείξει σήμερα μία λιγότερο αυστηρή στάση, να αλλάξουν τη στάση τους και να προστατεύσουν τις θάλασσές μας. Ευχαριστώ πολύ. Δύο λεπτά η κυρία Τίκαου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον συνάδελφο Ντεγκράντες Πασκουάλ για την προσπάθεια που έκανε. Πράγματι η μόλυνση στις θάλασσες είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε πολύ περισσότερο από όσο το κάνουμε. Ξέρετε ότι εμείς βιώνουμε το παράδειγμα της Μαύρης Θάλασσας. Η Μαύρη Θάλασσα τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί μια ιδιαίτερα μολυσμένη θάλασσα Υπάρχει υψηλή αζωτούχων, έχει δημιουργηθεί σοβαρότατο πρόβλημα και φυσικά και οι θαλάσσιες μεταφορές είναι υπεύθυνοι για το μεγαλύτερο ποσοστό της συγκεκριμένης μορφής μόλυνσης. Η συγκεκριμένη οδηγία ασχολείται με τις παράνομες απορρίψεις από πλευράς των πλοίων στη θάλασσα. Είναι αποτέλεσμα προσεξίας, αποτέλεσμα σκοπιμότητας μερικές φορές και θα πρέπει να εναρμονίσουμε καλύτερα τον ορισμό της ίδιας της ρήπανση από πλευράς των πλοίων και ε, να συζητήσουμε ακόμα περισσότερο τις κυρώσεις οι οποίες θα πρέπει να επιβάλλονται στα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Για να ενισχύσουμε λοιπόν και την θαλάσσια ασφάλεια και να μειώσουμε τη μόλυνση, έχουν ήδη γίνει ε, δεκτά ορισμένα μέτρα, το λεγόμενο πακέτο για τη θάλασσα, είναι κάτι το οποίο αφορά την εφοπλιστική οικογένεια, τις διάφορες χώρες, τον επιχειρηματικό κόσμο που ασχολείται με τις παράκτιες δραστηριότητες και με τις μεταφορές. Το σύστημα όμως έτσι όπως λειτουργεί σήμερα είναι θα έλεγα γραφειοκρατικό και επιβαρυντικό. Πάντως οι προτάσεις οι οποίες γίνονται είναι απαραίτητες και είναι απαραίτητες για τη σύμβαση Μαρπόλ η 73-78 δεν εφαρμόστηκε σωστά. Υπάρχει μια ελληματική εφαρμογή όλων αυτών των ρυθμίσεων. Γι' αυτό λοιπόν η ολοκλήρωση του πακέτου για τη θαλάσσια πολιτική είναι απαραίτητη και οι γνωμοδοτήσεις από τις διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές ήταν απαραίτητες. Η κυρία Λιούμπτσεβα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ Επίτροπε, ευχαριστώ συνάδελφοι. Είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο οφείλουν να προστατεύσουν τον Ευρωπαίο πολίτη ο οποίος πληρώνει το τίμημα της μόλυνσης των ακτών και των θαλασσών μας. Είναι προφανές επίσης ότι οι, ισχύουσα, οι ισχύουσες νομικές ρυθμίσεις δεν είναι επαρκείς και η εφαρμογή άλλωστε αυτών των ρυθμίσεων είναι ελιπεστάτη και δεν συνεισφέρει στη διατήρηση ενός καθαρού περιβάλλοντος των ακτών και των θαλασσών. Δεν αρκεί να έχουμε κανόνες, πρέπει να τους εφαρμόζουμε κιόλας. Θα πρέπει επίσης οι κυρώσεις για παράνομες απορρίψεις να μην είναι τόσο γελία, χαμηλές και είναι απαραίτητο να ενισχυθεί ο έλεγχος, να ενισχυθεί η επίβλεψη. Οι σύγχρονες τεχνολογίες μας διευκολύνουν προς την κατεύθυνση αυτή και θα πρέπει επιτέλους να σκεφτούμε ότι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι αναπόσπαστος στόχος μας και καθήκον μας. Και γι' αυτό είμαι υπέρ αυτής της αναθεωρημένης οδηγίας και είμαι υπέρ και της δημιουργίας του παρατηρητηρίου που θα ασχοληθεί με την εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων. Ευχαριστώ. Κύριε Ταγιάννη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμπερασματικά θα ήθελα να πω το εξής. Δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε την ευχαριστησή μας για τη διοργανική συνεργασία ανάμεσα στα τρία όργανα, όπως το υπογράμμισε άλλωστε και ο κύριος Γιαζεμπόσκη, ήταν ιδιαίτερα κακοφόρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για την προσπάθεια που έκανε Νομίζω ότι τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέδειξαν και στο τέλος αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου ότι είναι σε θέση να συνεργαστούν στενά και αποτελεσματικά και να καταλήγουν σε μία λύση και στην πρώτη ανάγνωση. Αυτό είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους Ευρωπαίους πολίτες. Ένα άλλο μήνυμα σημαντικό σε έναν τομέα τόσο σημαντικό όσο οι μεταφορές. Θέλω να ευχαριστήσω και την Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους ε, κοινοβουλευτικούς οι οποίοι συνεργάστηκαν με τις ομάδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πολλούς μήνες. Χάρης λοιπόν στην προσπάθεια όλων αυτών Αποδείξαμε ότι όταν μια γραφειοκρατική θα έλεγα δομή έχει συγκεκριμένους στόχους και μέσα δεν είναι σε καμία περίπτωση εμπόδιο η γραφειοκρατική αυτή δομή για τον πολίτη αλλά είναι κάτι το οποίο του διασφαλίζει σωστές λύσεις στα προβλήματά του. Ελπίζω αύριο το Κοινοβούλιο για μια ακόμη φορά να αποδείξει την αποτελεσματικότητά του και τη βούλησή του να στηρίζει πάντα τον Ευρωπαίο πολίτη με την ψηφοφορία το Συμβούλιο, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο καλύπτουν ένα νομικό κενό και θα επιτρέψουν από αύριο τα κράτη-μέλη να διώκουν σωστότερα αυτούς που μολύνουν τις θάλασσές μας. Μια επιπλέον ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση και την προστασία των δικαίων και των ελευθεριών του Ευρωπαίου πολίτη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. κύριε Ντεγκράντες λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε πολύ σύντομα και θα με ευχαριστήσετε που θα είμαι σύντομος. Θα ήθελα να πω το εκεί. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ για αυτά που είπατε. Όπως είπατε, η... το τρίτο πακέτο για την ασφάλεια της θάλασσας είναι πολύ σημαντικό και όπως αποδείχθηκε στο τέλος της θητείας αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να υπογραβήσουμε την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των κοινοτικών οργάνων, την ε, εξαιρετική συνεργασία που είχαμε με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τους και ηγητές. Πιστεύω τελικά ότι αύριο σε πρώτη ανάγνωση για ένα τόσο σημαντικό θέμα θα μπορέσουμε να ε, εγκρίνουμε την έκθεση που συμπληρώνει το ε, τρίτο πακέτο μέτρων για την ασφάλεια στις θάλασσες, πράγμα το οποίο είναι χρήσιμο, ε, επιτρέπει επικοδομητικό διάλογο υπέρ όλων και επιβεβαιώνει στα πλαίσια της απόφαση πόσο ε, σωστά γίνεται στην συνεργασία. Ευχαριστώ σας, ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε και ως πρώην του Κοινοβουλίου. Έληξε η συζήτηση, η ψηφοφορία της έκθεσης αυτής θα γίνει αύριο και τώρα συνεχίζουμε με την προφορική ερώτηση για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Πρώτος ηγητής, η κυρία Μακάρθη, για πέντε λεπτά. You seem